η Χιουρή ότι θα πρέπει να τιμούμε αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πρώτος και τώρα ε, ολοκληρώνεται εδώ πέρα η μονή της ομιλής και πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διατάξης, δηλαδή η έκθεση του κυρίου Αρσένη όσον αφορά την προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο εισηγητής. Commissioner, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας, για καθέναν που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, αλλά και για καθέναν Ευρωπαίο, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ευρώπης και αν βρίσκεται. Τα δάση είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας. Είναι η αναψυχή μας, είναι η απασχόλησή μας. Κι όμως τα δάση είναι τόσο διαφορετικά για το καθένα μας, την κάθε περιοχή της Ευρώπης αν κάποιος από την ε, βόρεια ευρώπη επισκεπτεί τα δάση της μεσογείου θα δει πολλά δάση που εμείς στη μεσόγειο θα ονομάζαμε δάση που θα τα θεωρούσε σαβάνα ή πάρκα καθώς δεν έχουν ε, παραγωγικές δραστηριότητες. ή αντίστοιχα κάποιος από τη μεσόγειο ταξιδεύει στη βόρεια ευρώπη θα θεωρήσει ότι τα δάση αυτά είναι πιο πολύ ανθρωπογενή παρά φυσικά καθώς έχουν πολύ έντονη την παραγωγική τους χρήση αυτά τα δάση που είναι τόσο διαφορετικά για καθένα μας ξεχωριστά στην ε, ευρώπη για κάθε μια περιοχή έχουν μια κοινή απειλή την κλιματική αλλαγή. η κλιματική αλλαγή απειλεί μέσα από την αύξηση των πυρκαγιών τις αρρώστιες που μεταδίδονται από ε, χώρα σε χώρα και απειλούν ολόκληρα είδη και άλλες καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα τα ευρωπαϊκά δάση. οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές ανά γεωγραφική περιοχή όμως είναι διασυνοριακές και απαιτείται η συνδρομή της Ευρώπης στην αντιμετώπιση τους. Σήμερα συζητάμε και σε δύο μέρες ψηφίζουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου για, την προστασία των δασών. Είναι μια έκθεση η οποία διαμορφώθηκε συνενετικά από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με βουλευτές από όλες τις χώρες και τα κόμματα και όταν κατατέθηκε στην προσέγγιση στην επιτροπή ακολούθησε μια διαδικασία 50 συμβιβαστικών τροπολογιών στη διαμόρφωση περαιτέρω της έκθεσης από όλε τι ε, κομματικέ παρατάξει και τι ε, περιοχέ ε, που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη. Γι' αυτό είμαι, νιώθω βέβαιο ότι αυτή η έκθεση εκπροσωπεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα δάση, να βοηθήσουν τις κοινωνίες μας να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή τι ζητάμε με αυτή την έκθεση. ζητάμε από την επιτροπή να προχωρήσει με τη λευκή βίβλο για την προσαρμογή των δασών για την προστασία των δασών στην κλιματική αλλαγή ζητάμε έναν νέο κανονισμό σε αντικατάσταση του παλαιότερου για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ζητάμε έναν νέο κανονισμό σε αντικατάσταση του παλαιότερου για την πληροφόρηση για τα δάση ζητάμε την αύξηση της χρηματοδότησης για τα δάση από τον πυλώνα 2 της κοινής αγροτικής μας πολιτικής. Τα δάση αντιπροσωπεύουν το 42% της υπαίθρου και όμως λαμβάνουν μόλις το 1% της ΚΑΠ. Ζητάμε να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης δημοσίων φορέων, να υπάρχουν κριτήρια βιωσιμότητας για, τα, τη διαστική βιομάζα που χρησιμοποιούμε για την ενέργεια και τέλος μια ενεργή ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών προσαρμοσμένη στην κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και ο πρώτος ομιλητής, η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπασέσκου. Η έκθεση αυτή θα ήθελε να προωθήσει την προστασία των δασών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασιζόμαστε λοιπόν στη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αρχών των κρατών μελών. Το άρθρο 203 μιλάει για την παράνομη υλοτομία. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Για να τεθεί σε αίσιο πέρας αυτή η διαδικασία, δεν θα πρέπει να υπάρχουν νομικά προσχώματα. Ως προς τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα ιδιαίτερα σε πολυμερές και διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα είναι ευρύτατο και θα ήθελα απλώς να εκθέσω δύο σκέψεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κινδύνους των ε, οικοσυστημάτων των δασών. Ιδιαίτερα τα εξωτικά είδη και οι πυρκαγιές. Αυτή Αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά, ιδιαίτερα στις χώρες του στόχου σύγκλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθετικότητα των δασών σε αυτά τα ε, βιωτικά και μη είδη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς έχει η φυτοϊγιεινή των δασών, λαμβάνοντας υπόψη την αναδάσωση και τα μεικτά δάση τα οποία είναι πιο ανθεκτικά. Δεύτερον, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στην μεγάλη διαφορά φυσικών ε, συνθήκων, μάλλον κλιματικών συνθήκων και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολυλειτουργικότητα των δασών μέσα στα πλαίσια της αγροτικής και μη ζωής. Ο κύριος Κέλλη. Όχι, ο κύριος Πάσκα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι πρόσφατες μελέτες για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών επί των δασών καταδεικνύει ότι τα οικοσυστήματα των δασών ε, αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα με την περίσταση και όλα εξαρτώνται από τις φυσικές συνθήκες μία συγκεκριμένη περιφέρειας για να δούμε πώς αντιδρά. Οι ορεινές περιοχές αντιδρούν διαφορετικά από άλλες περιφέρειες. Γι' αυτό όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται ως προς τις ε, κλιματικές αλλαγές. Για την Κεντρική Ευρώπη οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό περισσότερο από άλλες περιφέρειες. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ανθεκτικά και μη είδη. Θα πρέπει να έχουμε μία συγκεκριμένη θετική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιφερειών. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ήμουν στην Ιρλανδική Βουλή για να μιλήσω για αυτή την ιστορική ημέρα. Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη, ιδιαίτερα ως προς την κλιματική αλλαγή θα, πρέπει να μας απασχολήσει οι ανανεώσιμες, να μας απασχολήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να δημιουργηθεί ένα δάσος χρειάζεται πολύ καιρός. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει έρευνα για να δούμε πώς ε, οι απώλειες μπορούν να μειωθούν. Ένα σπίρτο μπορεί να απαλείψει χιλιάδες εκτάρια δασών. Γι' αυτό φτάνουμε σε μια διαδικασία αποψήλωσης. Θα πρέπει τα επόμενα έτη να αντιμετωπιστεί αυτό. Ελπίζω να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μελλοντικά. Ο Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ και θα ήθελα να πω στα αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου τώρα, τόσο αργά, τα εξή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Αρσένη για τις δεσμεύσεις και την εργασία του προετοιμάζοντας αυτή την έκθεση για την προστασία των δασών εν ώψη της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη για τη συνεισφορά τους. Σας είπα ότι θα υποβάλουμε μία, ένα πράσινο, μία πράσινη βίβλο για τις κλιματικές αλλαγές που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2010. Η πράσινη βίβλος που είχε ήδη υποβληθεί ασχολήθηκε με τα δάση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τις ε, δεκαετίες, τις επερχόμενες δεκαετίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι καλούμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν υπόψη ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στις εργασίες αυτές σε εθνικό επίπεδο και ανά την Ευρώπη. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι να αρκεστούμε στην αρχή της επικουρικότητας και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των δασών και οι πληροφορίες που έχουμε λάβει είναι διαθέσιμες. Πέρσι έγιναν πολλές συζητήσεις και μιλήσαμε και με τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να έχουμε μία διάδραση. Έγινε και μία σχηνοτενή συζήτηση για το κατά πόσο χρειαζόμαστε μία δασοκομική πολιτική ή όχι. Φαίνεται ότι το θέμα της δασοκομείας αποσχόλησε πολλούς φορείς, όπως διαφαίνεται και από την έκθεση που συνέταξε ο Κρήτον Αρσένης. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πληροφορίες για να δούμε θέματα ε, αποθεμάτων βιομάζας, γεών, βιοπικιλότητας, προστασίας των υδάτων και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να βρούμε μέσα για να το επιτύχουμε. Ήδη έχουμε αρχίσει τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και θα εργαστούμε και φέτος επί όλων των επιμέρους, επιμέρους ε, πτυχών που αφορούν τη δασοκομική πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε όλα αυτά τα θέματα που άπτονται και των περιβαλλοντικών και να έχουμε καλύτερο input έτσι ώστε τα δάση να μας ε, δίνουν πολλαπλά ευεργετήματα. Εμείς θα ε, εξετάσουμε αυτή την έκθεση και θα δώσουμε απαντήσεις και στους εμπλεκόμενους φορείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπη, σας ευχαριστώ συνάδελφοι που μείνατε τόσο αργά. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η συζήτηση έχει λήξει και η ψηφοφορία θα λάβει η χώρα την Τετάρτη. Η επόμενη συνεδρίαση θα, γίνει, θα αρχίσει αύριο στις